Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι πολύ καλύτερο μετά από τον κανονισμό αυτό, μετά την έγκριση του κανονισμού αυτού. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Σαΐε. Όταν μιλάτε για το ευρύ κοινό, ε, αναφέρεστε στον πρόεδρο φαντάζομαι, γιατί δεν έχουμε περισσότερο κοινό αυτή τη στιγμή. Και οι υπόλοιποι είστε υπερηδικοί, όλοι βουτυγμένοι σε αυτό το θέμα. Απολύτως και με πάθος λέγατε την άποψή σας περισσότερο λιγότερο συμφωνούσατε. Ολοκληρώνεται εδώ η συζήτηση. Αύριο θα γίνει η σχετική ψηφοφορία. Επόμενη συνεδρία της Ολομέλειας αύριο 5η, 16 Δεκεμβρίου. Είναι της Αγίας Αδελαίδας ε, των Καθολικών ε, και η μακαρίτησα η μητέρα μου λεγόταν Αδελαίδα. Έχετε λάβει την ημερήσια διάταξη και θα την βρείτε και στην ιστοσελίδα του Κοινοβουλίου. Λήξη συνεδρίαση μέχρι αύριο το πρωί. Και αύριο θα σας πω ε, χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα και ευτυχές στο νέο έτος, γιατί θα προεδρεύω και εγώ αύριο το πρωί. Καλό σας βράδυ, να είστε καλά.